So welcome everyone. Ξεκινάμε τη συστατική συντακτική ε, συνεδρίασή μας. Ο κ. Γκουέ αναπληρωτής Στίβεν Βούλφ, e είπαν ότι δεν το γνωστοποίησαν στη γραμματεία. Η δύο σε τέσσερα μέλη στην Επιτροπή. Έχει δικαίωμα η ομάδα να έχει τέσσερις ψήφους στη, στη απογευματινή συνεδρίαση. 16 μέλη έχουμε συνολικά που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Η γραμματεία έχει μάθει ότι θα συμμετάσχουν οι κάτωθοι αναπληρωτές που θα ψηφίσουν. ΕΛΚ. Αλέν Καντέκ, αντικαθιστά. Τον κύριο Ντάριος Ροζάτη, ΕΛΚ. Ο κύριο Αριζόφσκι, αντικαθιστά. Τον κύριο Γκούναρ Χόκμαν, Άλντε. Νίλ Στόρβαλτς, αντικαθιστά τον κύριο Μάικλ Τόιντερα, του Ρεσίνου. Μάικλ Ρέιμοντ, αντικαθιστά. Το μέλο μόλι Σκοτ Γκάτο, σοσιαλιστέ Τίμορ Σάντζι, αντικαθιστά τον κύριο Άλφρετ Σάντζο. Σοσιαλιστές. Ισαμπέλα Ντεμόντε αντικαθιστά τον κύριο Νάτο Σόρο. Φαντσουλίκα αντικαθιστά την κυρία Αμελής Ντότς. Προχωράμε τώρα. Θα εκλέξουμε πρόεδρο. Θα επαληθεύσουμε ότι έχουμε απαρτία. 15 μέλη που εκπροσωπούν τον τέταρτο των μελών της Επιτροπής. Είναι σαφές ότι έχουμε απαρτία. Εκλογή Προέδρου τώρα. Η κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του S&D προτείνω τον Ρομπέρτο Γκαλτιέρ να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εντάξει, δέχεται και ο Σγκουατιέρη να είναι υποψήφιος. Ο κύριος Γκαλτιέρη λοιπόν ανακηρύσσεται πρόεδρος της Επιτροπής. Και τον καλό να έρθει εδώ στο πρόεδριο. Thank you, Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Και το ευθύ αμέσω προχωρούμε στην εκλογή των αντιπρόεδρων. Οπότε τώρα, πέστε μα ποιοι είναι οι υποψήφοι για την πρώτη θέση αντιπρόεδρου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, σα συγχαίρω για την εκλογή σα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου να προτείνει τον συνάδελφο και φίλο Μάρκου Φέρμπερ. Thank Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλη υποψηφιότητα. Δέχεστε την υποψηφιότητά σας, μάλιστα. Now we can proceed. Και τώρα, συνεχίζουμε. Μπορείτε να προσέλθετε στα έδρανα του Προεδρείου. Yeah. Do I need Now Συνεχίζουμε τώρα για να εκλέξουμε τον δεύτερο αντιπρόεδρο, υποψηφιότητε. Φρέιρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Από πλευρά των Δημοκρατών προτείνουμε τον Πίτερ Σάιμον για τη θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου. Άλλε υποψηφιότητε. Δεν βλέπω. Άλλη υποψηφιότητα. Δέχεστε. All the candidates duly completed the declaration of financial interest. Όλοι οι υποψηφοί έχουν συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών ε, συμφερόντων και ο Μιλών και τώρα πάμε στο τρίτο αντιπρόεδρο. Υποψηφιότητε. Μάλιστα. Από πλευρά τη ομάδα ε, στήρικτων μεταρρυθμιστών προ τον κύριο Μπέρντ Λουκ. Άλλο υποψήφιο. Oui. Θα ήθελα να σας ζητήσω σύμφωνα με τον κανονισμό μας να γίνει μυστική ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη θέση. Ο πρόεδρος. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, και τουλάχιστον 10 να συμφωνήσουν με το αίτημα αυτό. Τουλάχιστον 10 θα πρέπει να συμφωνήσουν με το αίτημα. Yes. So now we have to proceed uh, on secret ballot election. That's... Προχωρούμε στην μυστική ψηφορία. Just a This, I first να σας πω ότι προβλέπει ο του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επομένως, θα πρέπει όλοι οι βουλευτές να έχουν την κάρτα ηλεκτρονική ψηφοφορία, να την έχουν έτοιμη και να την τοποθετήσουν στην σχισμή. Και μπορούν να ψηφίσουν ναι με το πράσινο κουμπί και όχι με το κόκκινο κουμπάκι. Σας αφήνω και το χρόνο, το ώστε να εξοικειωθείτε. Να συστηθώ, είμαι νέος. Θα ήθελα να συστηθώ, ρωτού ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είμαι νέος ευρωβουλευτής όπως είπα και θέλω να συστηθώ πρωτού ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ε, according to the uh, Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν προβλέπεται να γίνεται συζήτηση σε αυτού του είδους συνεδριάσεις. Σε αυτές τις συνεδριάσεις γίνεται μόνο η ψηφοφορία των Προέδρων και των Αντιπροέδρων. Οπότε με βάση τον κανονισμό θα γίνει η μυστική ψηφοφορία. Κυρία Φερέιρα παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε. Επειδή υπάρχουν πολλά νέα μέλη και επειδή θα γίνει μυστική ψηφοφορία, σας ζητώ να δοκιμάσουμε, να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα του ηλεκτρονικού συστήματος για να γνωρίζουν όλοι τι ακριβώς κάνουν κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας. Chairman, with your permission, on a procedural matter, my Για τα διαδικαστικά, ο κύριο Λόκα έχει ε, οριστεί ως υποψηφίος και ως, οι σοσιαλιστέ ζήτησαν να γίνει ψηφοφορία για το αν είναι καλό ή όχι. Νομίζω ότι είναι εντό του πνεύματο των κανονισμών να του δώσετε το λόγο για να εξηγήσετε για ποιο λόγο ε, θα είναι για ένας καλός υποψήφιος και το αντίθετο, αν δεν του το αφήσετε. Οπότε σα ζητώ να του δώσετε δύο λεπτά για να εκφωνήσει ένα μικρό λόγο για να μα εξηγήσει ποιο λόγο πρέπει να είναι αντιπρόεδρο. Ναι, μπορώ να δώσω τον λόγο. Κύριο Λούκα, δύο λεπτά το ανώτατο για να συστηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπέαντ Λούκε είναι το όνομά μου. Είμαι καθηγητής μακροοικονομίας πολιτικής οικονομίας δηλαδή με εξειδίκευση στην οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Εδώ και πολύ λίγο καιρό ασχολούμαι ενεργά με την πολιτική. Έχω εκλεγεί με το νέο κόμμα της Γερμανίας, την εναλλακτική για τη Γερμανία, διότι έχουμε μια κριτική στάση όσον αφορά την κρίση του ευρώ σε σύγκριση με τα άλλα γερμανικά κόμματα. Άκουσα τώρα ότι από την πλευρά κάποιων ομάδων υπάρχει η πρόθεση να μπλοκαριστεί η εκλογή μου. Γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω τον λόγο για να συστηθώ στους ε, συναδέλφους μου ώστε στο πλαίσιο της μυστικής ψηφοφορίας να μπορέσουν να λάβουν μια απόφαση. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο ε, ενδέχεται να υπάρξει αρνητική εκλογή ε, στην δική μου περίπτωση δεν αφορά προσωπικούς λόγους ούτε πιστεύω ότι υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τις ε, ικανότητες μου σε σχέση με την ε, οικονομική υποστήμη. Νομίζω ότι ο λόγος είναι η διαφορετική μου στάση όσον αφορά την κρίση του ευρώ από την πλειοψηφία των παρισταμένων. Θέλω λοιπόν να εξηγήσω τη θέση μου. Νομίζω ότι το ευρώ είναι ένα νόμισμα που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεγαλύτερη κρίση της ε, ύπαρξής της διότι τόσο όσον αφορά το δημόσιο χρέος όσο και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών δημιούργησε μεγάλες τάσεις και επιβαρύνσεις. Έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση αυτή μέσω ε, συνδυασμών ε, πολιτικών, συνδυασμού πολιτικών λιτότητας και μιας πολιτικής διευρυμένης ε, πιστοτικής ε, ε, απονομής πιστώσεων εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς με πολιτικές λιτότητας ο πρόεδρος ζητά να ολοκληρώσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Θεωρώ ότι η νεανική ενεργία και οι επιπτώσεις της λιτότητας συνιστούν επαρκή λόγο για να εξετάσει κανείς κριτικά την πολιτική για το ευρώ και τέλος θα ήθελα να ε, πω στους άλλους ευρωβουλευτές αν υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες ότι ε, βεβαίως θα σεβαστώ την εμπιστευτικότητα ε, πληροφοριών από πλευρά, παράδειγμα, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα και θα παραδίδεται τι ίδιε πληροφορίε στο Προεδρείο, όπω και όλα τα άλλα μέλη του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λούκε. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα, να δοκιμάσουμε πώ δουλεύουν οι κάρτε σα, πώ πάει όλη η διαδικασία. Κύριε Γκολάρη, διαδικαστικό. Ναι, να πω ότι είχαμε δικαίωμα κάναμε μάχες και σε αυτή την Επιτροπή ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία των φίλων μεταξύ των και αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει. Η γεωγραφική ποικιλομορφία είναι και σε αυτό σημαντικό επιχείρημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σταματάμε, δεν υπάρχει περιθώριο για συζητήσεις, δεν προβλέπει τον εσωτερικό κανονισμό, θα πρέπει να ψηφίσουμε, να δοκιμάσουμε πρώτα τα μηχανήματα και μετά να ψηφίσουμε. Ψηφίστε λοιπόν παρακαλώ. This is just a test. Δοκιμή είναι, έτσι. Δοκιμή. δοκιμή. Λοιπόν, μυστική δοκιμή θα κάνουμε. Ψηφίστε λοιπόν τώρα, μυστικά. Μυστικά. Δοκιμή μυστικής ψηφοφορίας. Δοκιμάζουμε το μηχάνημα. Are we having the right numbers? Να τσεκάρουμε, είναι σωστή αριθμή. E Ένας ΕΛΚ παραπάνω. Έχουμε μια ψήφο του ΕΛΚ παραπάνω. Εντάξει τώρα. One SD παραπάνω. Α βγάλει την κάρτα του ένα μέλο των σοσιαλιστών, παρακαλώ. Ένα μέλο του SND παραπάνω. I ask the socialist group. Η σοσιαλιστική ομάδα, παρακαλώ. Να φύγει ένα που περισσεύει. We have 17 SNDs. Έχουμε 17 και πρέπει να έχουμε 16 μέλη του SND. Δεν μετάτε τον πρόεδρο πιθανότατα. So, please, one of the substitute could... Ένας αναπληρωτής I asking the SND to cut one of the vote. Μία ψήφο βγάλτε παρακαλώ τα μέλη του SND. Yeah, this is there. Is there. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την πραγματική ψηφοφορία. Υπέρ. Αφήστε με να τελειώσω. Εκείνοι που υπέρ θα πατάνε πράσινο, εκείνοι που είναι κατά θα πατάνε το κόκκινο που μπει στο μηχάνημα. Αριστερά και δεξιά. Αριστερά είναι ναι, δεξιά είναι όχι. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay. We close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 30 ψήφοι κατά, 6 εποχές. Άρα, δεν εκλέγεται ο υποψήφιος. αναβολή εκλογής του Αντιπροέδρου για να δώσουμε χρόνο για προβληματισμό στις πολιτικές ομάδες. Όσον αφορά την ψηφοφορία για τον Αντιπρόεδρο, διακόπτεται η ψηφοφορία. Θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση, αρχές επόμενης συνεδρίασης, τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. δημοσίευση τη Δευτέρα.